υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Διοίκησης ε, της... Ε, η κυρία Ντελβό έχει πάλι το λόγο. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο αυτό ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετά χρόνια το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και ιδιαίτερα ακριβώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της αύξησης των υποθέσεων. Ο αριθμός των υποθέσεων αυξήθηκε από 398 το 2000 σε 12.000 το 2014. Οι υποθέσεις σωρεύονται από χρόνο σε χρόνο έχουν κατατεθεί επίσης και προσφυγές ε, για τις καθυστερήσεις. Ε, θεωρούνται παραβιάσεις των ανθρωπίνων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και υπολογίζεται αποζημίωση 27 εκατομμυρίων ευρώ, το διπλό του κόστους της μεταρρύθμισης δηλαδή. Γι' αυτό και ψηφίσαμε στις 28 Οκτωβρίου του 2015 υπέρ της προτάσεως του Συμβουλίου για την αύξηση των δικαστών στο δικαστήριο έτσι ώστε να είναι δύο δικαστές από κάθε χώρα να καταργηθεί το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης και να ενταχθούν οι δικαστές, οι δικαστές αυτοί στο πρωτοβάθμιο. Ο κανονισμός τον οποίο καλούμεθα να αποδεχθούμε είναι το δεύτερο στάδιο στην φάση αποδοχής μεταφορά δηλαδή των δικαστών, μεταφορά και όλων των υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς το κεντρικό δικαστήριο, στο γενικό καλύτερα δικαστήριο. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε στις μεταφορές αυτές ε, την ε, βεβαιότητα της δικαστικής διαδικασίας. Οι υποθέσεις λοιπόν θα συνεχίσουν να, να υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες. Ελπίζουμε ότι η αναδιοργάνωση αυτή θα προσθέσει ε, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στις εργασίες των δικαστών. Δεν θέλουμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας μόνο μια πιο γρήγορη απονομή, αλλά και μια ποιοτικότερη απονομή δικαιοσύνης. Ζητάμε λοιπόν έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται από τα διάφορα τμήματα του δικαστηρίου που αποτελούνται από πέντε δικαστές πλέον αντί για τρεις και ελπίζουμε επίσης από το δικαστήριο να υπάρξει διοργάνωση ειδικών τμήματων. Τονίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει επίσης στο εσωτερικό του δικαστηρίου ισότητα ανδρών γυναικών και υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά στα κράτη-μέλη να σεβασθούν τους διορισμούς. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η πρόταση η οποία γίνεται δεν είναι η καλύτερη. Λυπάμαι που τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για μια μικρότερη αύξηση του αριθμού των δικαστών και για ένα σύστημα εναλλαγής. Αλλά μπροστά στην έλλειψη ευελιξίας του Συμβουλίου εμείς αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δυσκολεύεται, πρέπει να την προστατεύσουμε δίδοντάς της τα μέσα να λειτουργήσει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα χώρο δικαιοσύνη στο εσωτερικό της Ένωσης, πράγμα κυρίαρχο στη δημοκρατία μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελβό. Είμαστε εν αναμονή της άφηξης του Επιτρόπου Αβραμόπουλου. Νάτος έρχεται. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ μπορούμε να ακούσουμε τη γνωμοδότηση της ε, Προέδρου της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων, της κυρίας ε, Γκέριγκεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας για πρώτη φορά οποιαδήποτε ε, μετατροπή του ε, καθεστώτος του Γενικού Δικαστηρίου θα πρέπει να γίνεται βάσει νομοθετικές διαδικασίες και η πρόταση που συζητούμε σήμερα είναι ε, για να αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες του Γενικού Δικαστηρίου και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος συνολικά με βιώσιμο τρόπο. Ε, πιστεύω ότι η έγκρισή του θα μειώσει τη διάρκεια των, της εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου και ε, έτσι να μην θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παραβιάζει τη συνθήκη θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπουν ότι πρέπει να εκδικάζονται υποθέσεις σε το χρόνο. Ε, Επίση, το δικαστήριο θα είναι υπεύθυνο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και να, θα πρέπει να ακούγονται όλες οι εφέσεις. Αυτό θα βολτιώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα και θα υπάρχει και συνέπεια στην ομολογία του δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την παρούσα πρόταση προκειμένου να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Σύστημα να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο, την κυρία Φιούμπνερ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Σας ε, παραχωρούμε ένα λεπτό. Ο Επίτροπος ζητά να παρέμβει εντός ολίγου, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ζιεύκα εκ μέρου του ΕΛΚ και, να ακούσουμε λοιπόν τι απόψει των ε, πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το δεύτερο στάδιο της μεταρρύθμισης του δικαστηρίου και πρόκειται για μια πολιτική συζήτηση αυτή που γίνεται εδώ για την ανάγκη διενέργειας της μεταρρύθμισης την οποία όμως ξεκινήσαμε πέρσι. Τώρα έχουμε την απαραίτητη συνέχεια αυτών που ήδη έχουν γίνει. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν το δικαστήριο στο γενικότερο δικαστήριο δεν θα είναι νέοι οι δικαστές, αλλά θα συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των δικαστών ε, στο υφιστάμενο όριο. Δεν υπάρχει έξτρα κόστος, δεν υπάρχουν επιπρόσθετες δαπάνες, υπάρχουν όμως επιπρόσθετα ωφέλη. Και οι δικαστές αυτές, αυτοί ασχολούνται κυρίως αποκλειστικά ε, με θέματα που άπτονται του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν τώρα να εμπλουτίσουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους και συνήθως ξέρετε δεν είναι πολλές οι εκκρεμείς οι υποθέσεις. Οι αλλαγές που έχουν γίνει θα μας επιτρέψουν οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν ε, το προσωπικό να δικάζονται στο πρωτοβάθμιο και άρα δεν υπάρχει ε, κανένας κίνδυνος. Θα εξεταστούν με τον δέοντα τρόπο ενώ οι δικαστές θα είναι σε θέση να ασχοληθούν και με άλλες υποθέσεις. Κάτι το οποίο ήταν ανέφικτο και αδύνατο μέχρι σήμερα. Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη και όπως είπε και η Ντανούτα Χιούμπνερ είναι μια μεταρρύθμιση που θα βελτιώσει την ποιότητα της, ε, του δικαστικού σκέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό το δικαστήριο και τα λοιπά θεσμικά όργανα να μην λησμονούν τη σημασία που έχει το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βέβαια θα αξιολογήσουν τη μεταρρύθμιση ενώ και άλλοι άνθρωποι και άλλοι φορείς που ενδεχομένως είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αξιολογήσουμε προσεκτικά τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγα χρόνια για να είμαστε σε θέση να πούμε ότι πράγματι κάναμε τη σωστή επιλογή. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, Ρέγναν ε, για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με αυτή τη μεταρρύθμιση, χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για μια τεχνική μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου και η συνέχεια στο, στο δικαστήριο Μαρίνιο όσον αφορά την αύξηση των μελών ώστε κάθε κράτος ε, μέλος να μπορεί να διορίζει δύο δίκαστες αυτό έγινε τότε υπό τους όρους ότι το δικαστήριο θα ε, διαλύεται όσον αφορά τις ε, δημόσιες ε, υπηρεσίες και οι ρυθμίσεις είναι τώρα σαφές, σαφέστερες και το τι ε, πρέπει να γίνει μια και δεν θα υπάρχει ειδικό δικαστήριο είναι σαφές. Με την τροποποίηση του οργανισμού, του μηχανισμού λειτουργίας ε, του δικαστηρίου είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και δεύτερον έχουμε ένα ξεχωριστό ε, ζήτημα εδώ που αποσαφηνίζει η έκθεση Ντελβό περισσότερο ότι μία ισόρυθμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και όσον αφορά τα αξιώματα των δικαστών πρέπει να διασφαλίζεται. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην ψήφιση της έκθεσης Μαρίνιο αυτό έγινε όρος και προϋπόθεση από εμάς και απευθύναμε έκκληση στο δικαστήριο να λάβουν υπόψη τους αυτή την ανάγκη όταν θα γίνονται διορισμοί και αυτό γίνεται επίσης και στο εθνικό επίπεδο ώστε να λειτουργεί η ισόρυθμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και αυτό επιθυμούμε να γίνεται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι, εξ ονόματος του ECR, παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, Συμφωνώ απόλυτα με την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήταν επιτέλους, ήρθε η χρονική στιγμή να συνταχθεί μια τέτοια έκθεση και να προχωρήσουμε. Βλέπουμε ότι υπήρχε ανάγκη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να συμβιβαστούν μεταξύ τους όλες οι πολιτικές ομάδες. Να μην ξεχνάμε και το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι αυτός ο συμβιβασμός μέσω της αύξησης του αριθμού των δικαστών μπόρεσε να επιτευχθεί. Θέλω να τονίσω κάτι, ότι αυτή η σημαντική τροποποίηση όσον αφορά την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 20 εκατομμύρια που συνεπάγεται αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύπτεται από πλευρά των Ευρωπαίων φορολογουμένων και των εισφορών τους. Και δεν υπάρχουν επαρκή τεκμήρια για μια τέτοια απόφαση που να δικαιολογείται με επιχειρήματα. Θα πρέπει λοιπόν από την άλλη πλευρά να λάβουμε υπόψη το κόστος σίγουρα πριν λαμβάνουμε οποιαδήποτε απόφαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιο Επίντο για δύο λεπτά εξ στον των Όπως λέμε στην Πορτογαλία, εκείνο το οποίο είναι στραβό από την αρχή δεν ισιώνει ποτέ. Και αυτό ήταν στραβό από την αρχή βλέπουμε. Η έλλειψη της διαφάνειας όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο ε, μας συνοδεύει χωρίς αμφιβολία και βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες καθυστερήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες. Εδώ και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υπήρξε βούληση από πλευράς του δικαστηρίου, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό και να μην ενημερώνεται όπως θα έπρεπε. Και έτσι λοιπόν να μην μπορούν να, να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι Ευρωβουλευτές. Όπως αναφέρεται στην έκθεσή μου, τα ειδικά δικαστήρια είναι πιο αποτελεσματικά και οι αποφάσεις τους είναι καλύτερης ποιότητας. Όμως υπάρχει αντίθετη επιλογή. Να υπάρχει δηλαδή εδώ μεγαλύτερη δαπάνη, μεγαλύτερη δισκαμψία και μεγαλύτερη δυσλειτουργία. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε ότι αποτελεί ένα ε, μεγάλο ψεύδος. Για το Γενικό Δικαστήριο οι εκκρεμότητες έπαψαν να, να υφίστανται, αλλά με τον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών, πράγμα που τεχνικά δημιουργείται μια κατάσταση υποαπασχόλησης για αυτούς και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν και οι νέοι δικαστές οι οποίοι θα διοριστούν να επιληφθούν περιπτώσεων. Ο αριθμός των υποθέσεων είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό των αποφάσεων προελαμβάνοντο. Και έχουμε και θέματα εδώ ε, μάρκας ε, και τα οποία αφορούν τον ε, ανταγωνισμό. Και βλέπουμε εδώ με προληπτική δράση της Επιτροπής έγινε αυτό. Το δικαστήριο το οποίο ομόφωνα αναγνωριζόταν για την εξαιρετική του νομική ποιότητα και είχε ένα δικαιολογημένο κόστος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από μια λύση η οποία φέρνει δαπάνες υπερβολικές εις βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων και μάλιστα χωρίς καμία δικαιολογία. Αυτό κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι μία από τις αρνητικές επιπτώσεις του σφάλματος που υπήρξε από την αρχή. Και έτσι το μέγιστο δαπανάτε για να έχουμε το ελάχιστο αποτέλεσμα. Δυστυχώς μία μέθοδος που πολύ συχνά ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Στρεβλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουτολα, εκ μέρου των Πρασίνων, για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η μεταφορά δικαιοδοσία σε διαφορέ ε, δημοσίων υπαλλήλων είναι μία από τι ουσιαστικέ αλλαγέ ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική να υπάρχει αγαστή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για όλη την νομοθεσία. Γι' αυτό και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουμε αποφάσει που ε, μπορεί και να προκαλέσουν πολλές επικρίσεις, αλλά παρόλα αυτά τις λαμβάνουμε. Μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου και τήρησε τις υποσχέσεις της προς το δικαστήριο και προς το Συμβούλιο. Και τα κράτη-μέλη όμως πρέπει να κάνουν και το ίδιο και αναφέρομαι και ε, σε αυτό. Ε, πέρσι υπήρχε ε, μια κοινή δήλωση που έλεγε ότι στο τέλος της διαδικασίας μεταρρύθμισης προκειμένου να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών τα κράτη-μέλη όσο το δυνατόν θα πρέπει να διορίσουν γυναίκες δικαστές για να υπάρχει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταλαντούχους και λαμπρούς δικαστές και άνδρες και γυναίκες και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το στο Συμβούλιο την υπόσχεσή του που φαίνεται να μην έχει τηρήσει μέχρι τούτε. Ευχαριστώ η κυρία Φεράρα εκ μέρους του EFTD για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στην ε, πολλωστή πράξη που όπως και η ίδια η συγγήτρια η κυρία Ντεβελβό ε, χαρακτήρισε μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, ή εγκρίναμε το διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών ε, και περάσαμε από τους 28 στους 56 δικαστές για το Γενικό Δικαστήριο. Τώρα το Κοινοβούλιο θέλει να εγκρίνει την κατάργηση του ε, Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, μία απόφαση όπου το θέμα της συνταγματικότητας αμφισβητήθηκε από νομικούς, από πανεπιστημιακούς και από το ίδιο το δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Πιστεύω ότι όσον αφορά την κατασπετάληση των δημοσίων πόρων, ε, όσον αφορά τις εγγυήσει για τη μετερρύθμιση, μας φαίνεται πάρα πολύ αμφισβητήσιμο ότι είναι στη δικαιοδοσία του νομοθέτη να δημιουργήσει και άλλα δικαστήρια και επίσης να αποφασίσει την κατάργησή τους, δημιουργώντας μία αρχιτεκτονική δικαστική δομή που σίγουρα ε, έχει συνταγματικά προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε στο κράτος δικαίου και επομένω δεν μπορούμε να εγκρίνουμε με μεταρρύθμιση που παραγνωρίζει τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάγερ για την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα δικαστήρια και οι διαδικασίες τους, οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι ο πυρήνας της ε, νομολογίας και πάντα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και όλο και περισσότερο όταν πρόκειται για τη σύνθεση των δικαστηρίων και όταν εμπλέκονται πολιτικοί εδώ και οι πολιτικοί και οι πολιτικοί άνδρες. Εδώ υπάρχει δικαίωμα για ταχεία λήψη αποφάσεων και σύντομες διεργασίες, διαδικασίες και για τις δαπάνες ε, από πλευράς δικαστικού κόστους ε, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία τελευταία χρόνια σημαντικά. Λοιπόν, όσον αφορά την, την σύνθεση των δικαστηρίων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι διεργασίες όμως είναι εκείνες ε, που με ενοχλούν και είναι μια, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήθηκαν 12 ε, πρόσθετοι δικαστές ε, και τι γίνεται τώρα, 28 διορίζονται συνολικά. Διαρωτώ με τι γίνεται με τους 16 δικαστές που δεν τους χρειαζόμαστε. Θα κάνουν περιπάτους και ποιος θα πληρώνει αυτή την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς ε, οδηγούν στο να χωλένουν τα πράγματα στο τέλος τέλος ε, με τέτοια προβλήματα. Και εκείνο το οποίο με απασχολεί είναι οι δεξιότητες ε, των δικαστών αυτών όταν βλέπουμε ότι πολιτικά διορίζονται. Ευχαριστώ. Η κυρία Σταρά Φεραγούτ, αλλά δεν τη βλέπω εδώ στην αίθουσα. Επομένω μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Κοφεράτη, για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πριν από κάποιους μήνες εξέφρασα εδώ στην σχετική συζήτηση την αντίθεσή μου ε, για το διπλασιασμό των δικαστών για λόγους που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε κάποια θεμελίωση, δεν είχε κάτι λόγο να ψηφιστεί και ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει ε, μια περαιτέρω αποδιάρθρωση μιας δομής που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα όσα έχει κάνει η κυρία Ντελβό είναι πάρα πολύ σημαντικά προσπαθεί να διορθώσει κάποια από τα στρεβλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ εύκολα προβλέψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πλέον να φροντίσουμε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα το απορροφήσει το υπόλοιπο δικαστήριο και το οποίο στα ε, πλαίσια των ετών ε, ορίμασε με πάρα πολύ πολύτιμες αρμοδιότητες να μην χάσει αυτές τις αρμοδιότητες γιατί αν γίνει αυτό ε, πέραν της ζημίας θα έχουμε και το φταίξιμο. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το οποίο επενθυμίζεται πανηλημένως, η αναγνώριση των γυναικών σε αυτή τη δραστηριότητα, τη ισότητα δηλαδή μεταξύ των φίλων στη λειτουργία του μελλοντικού δικαστηρίου. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, χρειάζονται δεσμεύσεις. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ε, ε, αξία της γυναικείας εργασίας, την παρουσία των γυναικών, αλλά δεν θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν το θέμα αυτό απλώς το επικαλούμαστε και δεν μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις, πιστεύω ότι θα χάσει αξία και αξιοπιστία ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δεσμευτικές ποσοστώσεις και να εισαχθούν για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο κανόνας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοφεράτη. Ε, ο κύριος Ουγιαζτόφσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η απορρόφηση του ε, Δικαστηρίου Γενικών Αρμοδιοτήτων ε, των υποθέσεων δημόσιας διοίκησης από το Γενικό Δικαστήριο αποτελεί μήμα ενός ε, σχεδίου, ευρύτερου σχεδίου και σε αυτή την πολύ σύντομη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και κάποιο χρόνο τώρα, καταδεικνύεται το ότι πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο για τα μεθοδολογικά θέματα της υλοποίηση της ε, δικαστικής μεταρρύθμισης. Πολλά επιχειρήματα προαναφέρθηκαν όσον αφορά τις επικρίσεις ε, που έχουν ε, εγερθεί κατά της μεταρρύθμισης αυτής και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι οι ίδιοι οι δικαστές ε, ε, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που οδηγεί στο να συζητούμε το κόστος ε, της μεταρρύθμισης και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσα στο πλαίσιο της συνολικής συζήτησης για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον ανοιχτό του χαρακτήρα, αποτελεσματικότητα και ε, διαφάνεια των ε, αποφάσεων στην νομολογία. Και από πλευρά τώρα των όσων ακούσαμε, εγώ θα επέλεγα για ε, μια άλλη σκέψη που θα έπρεπε να μας ε, διέπει και να μας οδηγήσει προτού αποφασίσουμε στο τέλος τέλος το τι θα κάνουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και δεν είναι δυνατόν ε, ελαφρά την καρδία βιαστικά να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Μπουτονέ για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φτάνουμε στο τέλος της τέταρτης μεταρρύθμισης του δικαστηρίου με την κατάρχηση της δυνατότητάς του να δικάσει σε πρώτο βαθμό τις διαφορές μεταξύ των υπαλλήλων. Ε, με σκανδαλώδη τρόπο έγιναν όλα αυτά, δεν έγιναν με σωστή ανάλυση της νομικής βάσης, δεν έγινε ανάλυση αξιολόγησης αντικτύπου, του κόστους, αλλά ούτε ανάλυση για τις συνέπειες στα άλλα δικαιοδοτικά όργανα. Και αυτό επανειλημμένως το υπενθυμίσα στις διάφορες επιτροπές. Συνεχώς γίνεται λόγος για το πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο ενώ οι χώρες πλήττονται από τη λιτότητα. Και είδαμε ότι δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους ε, δημοσίους λειτουργούς ούτε με τους δικαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίστε έτσι και θα συνεχίσετε να αποκαλύπτετε το φρικτό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό δεν είναι η πτώση αλλά η προσγείωση και η δική σας κατάρρευση ε, πλησιάζει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπισιλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι το φθινόπωρο συζητήσαμε τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου και τότε είπα ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών. Είναι πολιτική απόφαση και δεν την υπερψήφισα. Σαφέστατα η ατζέντα του δικαστηρίου όλο και μεγαλώνει, αλλά δεν αρκεί για να ε, δικαιολογήσει την αύξηση ε, του αριθμού των δικαστών από 28 σε 56. Είναι ε, βεβαίως ο φόρτος εργασίας μεγάλος, αλλά δεν είναι δυνατό να έχουμε τέτοια αύξηση. Στην Τσεχία ε, Επίση, υπάρχει μεγάλος φόρτος στα δικαστήρια. Θα δεχόμασταν μια μικρή αύξηση του αριθμού ε, δικαστών, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση... Μάλλον είναι καλό πράγμα το ότι καταργήθηκε το πρώτο δικαστήριο και ενσωματώθηκε στο γενικό δικαστήριο. Θα έπρεπε να είχαν βρεθεί ε, τρόποι εξοικονόμησης των δαπανών. Νομίζω ότι έχει γίνει, έχει γίνει λάθος ο... οργάνωση της μεταρρύθμισης. Ίσως οι δαπάνες του αριθμού των δικαστών αντισταθμιστούν από τη μείωση των εξόδων λειτουργίας. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με την μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων. Δυστυχώς όμως πρόκειται για μια πολιτική μεταρρύθμιση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην κοινή λογική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε τώρα τη διαδικασία του Catch the Eye. Ο κύριος Νεγκρέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι το κόστος είναι το πρόβλημα. Το τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το δικαστήριο είναι το πρόβλημα. Ε, με την μεταρρύθμιση αυτή βελτιώνεται η κατάσταση. Άλλωστε ο κανονισμός αυτός είναι το προϊόν διαθεσμικού διαλόγου και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε μόνο τους διαδικαστικούς κανόνες ε, του δικαστηρίου, αλλά και άλλα πράγματα. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανεμηθεί και να διανεμηθεί ένας πιο μεγάλος αριθμός υποθέσεων όταν αυτό το επιτάσσει η σημασία των υποθέσεων αυτών. Μπορούν να γίνουν συνέργειες και θα πρέπει να ε, προσαρμοστούμε στις εξελίξεις. Τέλος, θα πρέπει να τηρηθούν τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί όλες αυτές οι αποφάσεις συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Πρόεδρε, συζητούμε για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της. Αρχικά είχε προταθεί από το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου σε 56, ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ορίζει από δύο δικαστές παράλληλα η αύξηση αυτή προϋπέθεται και την κατάργηση του δικαστηρίου δημόσιας διοίκησης. ωστόσο με τον παρόντα κανονισμό αυτό που αποφασίζεται είναι η αύξηση του αριθμού των δικαστών του γενικού δικαστηρίου από 40 σε 47 καθώς επίσης και η κατάργηση του δικαστηρίου της δημόσιας διοίκησης που αποτελείται από 7 δικαστές που θα μεταφερθούν στο γενικό δικαστήριο. τέλος δεδομένου ότι μεταξύ του 2000 και 2010 υπήρξε αύξηση κατά 65% των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο γενικό δικαστήριο ενώ στο τέλος του 2010 εκκρεμούσαν 1.300 υποθέσεις, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών σε 56, δύο ανά κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας στο Γενικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος ε, Παρακαλώ, Eh, Ευχαριστώ. Η συνεκτικότητα, στη συνέχεια, η προστασία, νομική προστασία των πολιτών, η αποτελεσματικότητα, όλα αυτά είναι αρχές και αξίες που αναφέρονται στην έκθεση και θέλω να πω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, για κάποια ζητήματα. Δεν έχω τη βεβαιότητα ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα οδηγούσε στα αποτελέσματα που επιθυμούμε και δεν γνωρίζω ότι δεν, είμαι καθό... δεν υπα... έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν σημαντικά λοιπόν θέματα που πρέπει να εξεταστούν και σοβαρέ προτάσει που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είμαι υπέρ τη μεταρρύθμιση, αλλά πρέπει σταδιακά, βήμα προ βήμα να υλοποιηθεί. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε, να βρούμε τον εαυτό μα όπου η έκθεση αυτή θα υποστεί σοβαρότατε επικρίσει. Είμαι υπέρ τη μεταρρύθμιση, αλλά βήμα προ βήμα, σταδιακά κλίμακοτα και αν θέλουμε πραγματικά να υιοθετηθεί η απόφαση ότι θα υπάρχουν δύο δικαστές κράτος μέλος τότε θα πρέπει η αρχή της ισότητας και αναλογικότητας να γίνεται σεβαστή. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ και η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Αβραμόπουλο που παρακολούθησε όλη τη συζήτηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να παρέμβει σε αυτή τη συζήτηση, η οποία, όπως επανέλαβαν αρκετές φορέ, βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Ντελβό. Παρακαλώ, Μάντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλα σε αυτή τη συζήτηση. Είναι η δεύτερη φορά σε έξι μήνες που το συζητούμε. Οι θέσει των ΜΕΝ και των ΔΕ δεν έχουν αλλάξει. Επομένως, ε, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ε, ότι ε, έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τη δικαιοσύνη, όλα τα δικαστήρια, αλλά κυρίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είμαι βέβαιη ότι θα οργανωθεί καλύτερα εάν οργανωθεί το ίδιο στην υπηρεσία της δικαιοσύνης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά στα κράτη-μέλη να ε, φροντίσουν να διορίσουν και γυναίκες ε, ώστε να υπάρχει ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελβό. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το